είναι η σειρά που προβαδίσματος που ακολουθείτε μετά την ε, εκλογή τους. Σας λέω λοιπόν τα αποτελέσματα με τη σειρά των ψήφων. 672 ψήφοι. 17 άκυρες ψήφοι. Έγκυρα ψηφοδέλτια 655. Έλαβον Ζωάννη Πιτέλα, 319 ψήφους. Μικέλ Άγχελ Ματίνες, 295. Άννη Ποδηματά, 281. 281 ψήφους. Αλέχο Βιδαλ 269 Γεώργιος Παπαστάμκος 248 Ρομπέρτα Αντζελίλη 246 Ότμαρ Κάρα, 244 Έντουαρτ Μακμίλαν Σκότ 239 Ιζαμπέλ Ντυρό. 238. Αλεξάνδρ Άλβαρο. 235. Ράινερ Βίλαντ. 230. Όλτριχ Φλάσακ, 223. Ε, Γιάσεκ Ποσαζιέβιτς. 206. Και Λάσλο Σουριάν. 188. Όλοι οι υποψήφοι λοιπόν έχουν εκλεγεί και μπορούν λοιπόν να θεωρηθούν ως εκλεγμένοι αντιπρόεδροι. Θα ήθελα να ξέρω αν κάποιος δεν δέχεται την εκλογή του στο αξίωμα του αντιπρόεδρου μεταξύ των υποψηφίων, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μπορώ λοιπόν να συγχαρώ όλους τους εκλεγμένους αντιπροέδρους. Κυρίες και κύριοι, η σύσταση του Προεδρείου είναι δεδομένη λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει στη συνέχεια η σειρά των συγχαρητήριων και τώρα θέλω να δώσω το λόγο αμέσως στον πρόεδρο Μπαρόζο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύρια Πρωθυπουργέ Θόνινγκ Σμιτ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω κυρία Πρωθυπουργέ για